Chers collègues, nous allons reprendre. Nous sommes déjà un petit peu en retard. Merci. Euh. Να συνεχίσουμε γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω και όποιοι θέλετε να μιλήσετε παρακαλώ έξω από την αίθουσα. Δεν λέω, το καταλαβαίνω ότι θέλετε να μιλήσετε, αλλά ενοχλούνται όσοι είναι εδώ. Να καλωσορίσω τώρα τους ε, προσκεκλημένους μας. ανησυχεί η διεθνής κοινότητα. Παρακαλώ. Καλωσορίζω λοιπόν τους προσκεκλημένους μας και ταυτόχρονα πρέπει να φωνάζω γιατί δεν κάνει τη ησυχία. Αφού καλωσορίζω από την ΕΕΔ και τον κύριο Ταπαταμπάη, λοιπόν να πω ότι υπάρχει αυτό το ψήφισμα που λέει ότι δεν σέβεται το Ιράν τη συμφωνία. Υπάρχουν επτά ψηφίσματα του ΕΕ που ζητούν από την Χεράνη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα και επιβάλλει κυρώσεις. Στο Ιράν ε, το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015 μεταξύ Ιράν, Κίνας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ρωσίας, Ηνωμένου Βασιλείου και είπα σημαντική πρόοδος που ε, βοηθάει τη μη διάδοση, περιλαμβάνει κάποιες διατάξεις με αντάλλαγμα την άρση ε, των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί.

που μπορεί να επιτρέψει στα 10 χρόνια τα επόμενα να πανευθούν οι κυρώσεις. Οι ανακοίνωσαν ότι προτίθεται να αποχωρήσουν από τη συμφωνία το 18 και έχουμε τις ε, τρεις ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, που θέλουν το αδιέξοδο να λυθεί μέσω επικοδομητικού διπλωματικού διάλογου. Από τον Ιούνιο βλέπουμε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση ε, της έντασης με τη ΣΥΠΑ. Ο πρόεδρος ε, του Ιράν είπε ότι δεν θα σεβαστεί πλέον τους περιορισμούς της Συμφωνίας του 2015. Το Ιράν δεν έχει αυξήσει τα επίπεδα ε, εμπλουτισμού ουρανίου μέχρι στιγμή. Αφήνει αυτό ανοιχτή την πόρτα σε μια διπλωματική λύση. Γαλλία, Γερμανία, Ενωμένο Βασίλειο ζητούν από το Ιράν να σεβαστεί τις υποχρεώσεις και είπαν ότι προτίθενται να ομολογήσουν το μηχανισμό επίλυσης ε, διαφορών. Υπάρχει δύο μήνες ε, διορία για διαπραγματεύσεις. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα λεπτή και τεταμένη με πολλούς κινδύνους. Θα τα πούμε όλα αυτά σήμερα. Έγινε και μια επίσκεψη πρόσφατα στο Ιράν για την επίλυση του αδιεξόδου. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Βυσσισικόφσκι, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ΑΦΚ και μετά του δύο προσκεκλημένου μα από την ΕΔ και τον κύριο Ταπαταμπάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που κάνετε αυτή την ε, συνεδρίαση. Την Υποεπιτροπή. Ε, πρέπει να συζητήσουμε το καθεστώς της συμφωνίας για τα πυρηνικά με το Ιράν και την ε, συμμόρφωση του Ιράν. Η συμφωνία με το Ιράν, το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση, ε, είναι προς το κοινό μα συμφέρον, είναι μέγιστο επίτευγμα για την περιφερειακή ασφάλεια και θέλει να αποτρέψει τον, την κούρσα για τα πυρηνικά. Οι πρόσφατε εξελίξεις στην περιοχή, ο θάνατος του στρατηγού Σουλεϊμανή, μας υπενθυμίζει τη σημασία της αποτροπής ε, καταστροφικών περιφερειακών σειράξεων και η αποκλιμάκωση είναι πολύ επίκαιρη σήμερα, πολύ περισσότερο από ποτέ. 21 Φεβρουαρίου Παρασκευή το Ιράν θα κάνει την 11η ε, κοινοβουλευτική, τις 11 κοινοβουλευτικές εκλογές της. Πολλοί αναλυτές προβλέπουν ότι η σκληροπυρηνική ε, θα κερδίσουν στο Κοινοβούλιο. Οι μεταρρυθμιστές ε, και οι μετριοπαθείς ε, υποψήφοι που το Συμβούλιο των Φρουρών τους αποδυνάμωσε, αποδυναμώθηκαν ακόμα περισσότερο μετά την απόφαση των Αμερικανών να, να αποχωρήσουν από την συμφωνία του 18 και τον κίνδυνο των κυρώσεων. Μία σειρά από ε, ψηφίσματα έχουν ε, υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ζητά το ΟΗΕ να σεβαστεί το Ιράν τις υποχρεώσεις του. Ε, θέλουμε μια πολιτική λύση λόγω των, της κλιμάκωσης. Επομένως, Πρόεδρε, ε, πρέπει να συζητήσουμε το μηχανισμό επίλυση των διαφορών και να το συζητήσουμε πολύ συνεκτικά. Ο Χασάν Ρουχανί, ο Πρόεδρος, ε, το γεγονός ότι η Ευρώπη κατά την άποψή του, έχει προβεί σε μία απόφαση που δεν συνάδει με το άρθρο 36 της Συμφωνίας ε, για τα πυρηνικά με το Ιράν. Πρέπει να αποφύγουμε την κατάσταση του μπαστούνιου και του καρότου, αυτής πολιτικής που ήταν αυτή που δέσποζε στο τοπίο προς της συμφωνίας με το Ιράν. Ε, θα σταματήσω εδώ. Ε, θέλω να ακούσω τα σχόλια. Είμαι πρώην πρέσβης της Πολωνία στο Ιράν και άρα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ε, θέλω να ακούσω τα σχόλια και τις απόψεις των δύο ομιλητών, των δύο βασικών ομιλητών του πάνελ για το θέμα αυτό. Σας δίνω και τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα δώσω το λόγο στον Μπρούνο Σόλτα, εκπρόσωπο της ε, ΕΣΕΑΕ. Ε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε την αποψή του για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνει ούτω ώστε να κάνει το Ιράν να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του προς την συμφωνία και να επιβιώσει αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και που θέσατε το πλαίσιο και τονίσατε και την ευαισθησία της κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει και για τη συμφωνία με το Ιράκ. Uh, e πω αυτής εξ εξαρχή, uh, ότι είμαστε δεσμευμένοι να κάνουμε πάνω δυνατόν ώστε να διατηρηθεί το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά διπλωματική ε, στο επίπεδο αυτό. Είναι όμως πιο ευρύ λίγο το πεδίο της συζήτησης. Θα μιλήσω για τη συμφωνία για τις εγγυήσεις, το, προ, το πρωτόκολλο και τη διάθεση για τη μη, μάλλον τη για τη μη διάθεση και μετά θα περάσω στο καινούργιο σχέδιο δράσης, τη συμφωνία με το Ιράν δηλαδή. Όλα αυτά πάντα από το πρίσμα αυτή το σχέδιο. Σε ό,τι αφορά τις ιρανικές ε, υποχρεώσεις ε, πρέπει να πω ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία ε, σε, ήδη από το 1973 με τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, δικαιώματα πρόσβαση και υπεγράφηκε ένα το πρωτόκολλο το 2003, πιο σημαντικό αυτό, διότι δίνει ευρύτερη πρόσβαση, σημαντικά ευρύτερη πρόσβαση σε πυρηνικό υλικό, σε καταστάσεις ε, και όλα τα εχέγγυα, όλε οι εγγύσεις και οι σχετικέ πληροφορίες παρέχονται. Ε, η Διεθνή Επιτροπή Ατομική Ενέργεια μπορεί να έχει πρόσβαση μέσα μετά από κοινοποίηση ε, προ δύο, δύο ωρών δύο ώρες νωρίτερα, να επισκεφθεί και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα Ιράν. Το 2003 όμως τότε δεν είχε επικυρώσει αυτό το, το πρωτόκολλο, αλλά μόλις το 2015 το έκανε στο πλαίσιο των δεσμεύσεών του σε αυτό το κοινό οργανωμένο σχέδιο δράση, όπου και δεσμεύτηκε ότι προσωρινά θα εφαρμόσει το πρόσθετο πρωτόκολλο. Και αυτό το λέω απλά για να υπογραμμίσω ότι εάν χαθεί αυτό, αυτή η συμφωνία χάνονται και όλα τα πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης δυνάμει του πρόσθετου πρωτοκόλου. Και αυτό θα είναι κάτι σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιολόγηση της ε, συμμόρφωσης του Ιράν της δεσμεύσει του, στην Ένωση εμείς βασιζόμαστε βέβαια στην Εθνική Επιτροπή των Κοινωνίας που είναι αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των σχετικών θεμάτων ε, όπως κάνει ήδη ε, εδώ και 60 χρόνια και ήδη από το 2013 έχει κάνει πολλές ε, εκθέσεις και από το 2015 και μετά για την υλοποίηση της Συμφωνίας περί και του πρόσθετου Πορτοκόλου. Από το 2015 η Διεθνής Επιτροπή στις αναφορές της ξεκάθαρα λέει ε, ότι συνεχίζει να επαληθεύει η τιμή μετατροπή έχει πρόσβαση, ε, μάλλον την ανάγκη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις. Τα λέει αυτά σε εκθέσεις που είναι δημόσιες, προσβάσιμες από τον ε, ιστότοπο της, στο Ιράν δηλαδή. Μέχρι στιγμής εφαρμόζει τη συμφωνία και το προς το πρωτόκολλο και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Και τώρα έρχομαι στο κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση, όπου εδώ η εικόνα δεν είναι και τόσο απλή, είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Στο πλαίσιο αυτού τη συμφωνία, το Ιράν ανέλαβε πρόσθετε εθελοντικέ δεσμεύσει ε, που δεν καλύπτονται από την προηγούμενη συμφωνία για τη διάδοση και το έκανε με αντάλλαγμα, πρέπει να το πούμε, την άρση των κυρώσεων. Όλοι τα ξέρουμε, 12 χρόνια χρειάστηκε η διαπραγμάτευση συμφωνία, την οποία έκρινε με ψήφισμα το 2231. Ε, συγκεκριμένα το Συμβούλιο Ασφαλείας, σημαντική επιτυχία και πρέπει να διατηρηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας τα δύο τρίτα των ε, μηχανημάτων ε, φυγοκέντρησης ε, τα ε, αποσυναρμολόγησε το Ιράν, πήρε και άλλα μέτρα μετά από την υλοποίηση ε, των δεσμεύσεων το 2016 ε, εφάρμοσε για τρία χρόνια ε, τις δεσμεύσεις του και μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ και την επαναφορά κυρώσεων. Είναι λυπηρό το ότι έχει συμβεί, το έχουμε πει το Μάιο το Ιράν ανακοίνωσε όμως ότι περιοδικά θα πάψει να εφαρμόζει τις δεσμεύσεις του λέγοντας ότι οικονομικά δεν έχει υποφεληθεί από την άρση των κύρος. Το λεγόμενο less for less. Αυτή η προσέγγιση λιγότερα για λιγότερα είναι μια προσέγγιση βέβαια που εμείς ποτέ δεν έχουμε δεχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον Ιούλιο του 2019 το Ιράν έχει κάνει τέσσερα βήματα για τη μείωση της αφαρμογής των δεσμεύσεών του. Το πρώτο βήμα ήταν σε ό,τι αφορά το επίπεδο εμπλουτισμού του ε, ουρανίου και τις ε, δραστηριότητες έρευνας ε, και ανάπτυξης έχει ξεκινήσει υπόγειες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του ουρανίου. όλα αυτά τα έχει διαπιστώσει και τεκμηριώσει και η Επιτροπή τον Γενάρη. το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει και σε ένα πέμπτο βήμα μείωση των δεσμεύσεων ε, τα επιχρησιακά όρια θεωρεί ότι δεν δεσμεύεται πλέον από αυτά και, και αυτό είναι σημαντικό. Να πούμε ότι είμαστε σε συνεχή επαφή με τη Διεθνή Επιτροπή των ενέργεια. παρακολουθούμε και τις αναφορές της μέχρι στιγμής, όμως δεν έχει εφαρμόσει το πέμπτο αυτό μέτρο το Ιράν που υποτείνει και το τελευταίο. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι κάτι τέτοιο είναι θετικό, γιατί όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά. Είπατε εκπρόσωπος και οι προηγούμενοι και τώρα, κ. Μπορέλ, έχουν εκφράσει την ασχέα. του, ζητούν πλήρη εφαρμογή, δεν θέλουν το less for less. Ταυτόχρονα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι σημαντικό να παραμείνει σύμφωνα με το Ιράν, γιατί υπάρχουν διατάξεις σε σχέση με την πρόσβαση. Είπα και το πρόστο πρωτόκολλο πριν. Αλλά και τον εμπλωτισμό του πλουτονίου, ε, αντιδραστήρα Σάρα κτλ. Υπάρχουν δεσμεύσεις, ε, πρέπει να τηρούνται. Και σε ό,τι αφορά το feedback που είχαμε από την Διεθνή Επιτροπή, έχει πει το Ιράν και το πράτη ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται και να παρέχει πρόσβαση στη Διεθνή Επιτροπή. Στοιχεία σημαντικά και αυτά που δείχνουν ότι ακόμα δεν έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, κάποιες τελευταίες ε, εξελίξεις, περισσότερες, πιο οξυμένες περιφερειακές εντάσεις και 14 Ιανουαρίου, επιπροσθέτως, ε, η Υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου ενεργοποίησαν τον μηχανισμό ουσιαστικά επίλυσης ε, διαφορών λόγω των βημάτων που έχει κάνει το Ιράν για περιορισμό των δεσμεύσεών του. Με την ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού βέβαια ξεκαθάρισαν ότι αυτό το κάνουν με βασικό σαφή στόχο την επίλυση ε, της διένεξης. Κάποιες φορές παρουσιάζεται λάθος ως ένα ε, μέτρο κλιμάκωσης. Το είπαν και δημοσία ότι ο στόχος τους είναι να ε, λυθούν τα ζητήματα που εκκρεμούν. Ο υπάτος εκπρόσωπος, ο συντονιστής και η Διεθνή Επιτροπή των Ανάγκη σε διαφορετικά επίπεδα δραστηριοποιήθηκαν στη στενή επαφή με όλου του συμμετέχοντε σε αυτό το κοινό σχέδιο δράση. Ο υπάτος εκπρόσωπος πήγε στο Ιράν, μίλησε και επίσης με τους Κινέζους Ρώσους ομολόγους και μετά από διαβουλεύσεις αποφασίστηκε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες και η διαδικασία ε, θα παραταθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συνομιλίες ε, σε επίπεδο ειδικών μεταξύ όλων των συμμετέχοντων σε αυτό το κοινό σχέδιο δράσης για να διασκεδαστούν οι πυρηνικέ ανησυχίε και να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερε επιπτώσει αποχώρηση των ΗΠΑ συμφωνία και τη ε, επανεπιβολή κυρώσεων. Επίση, το Ιράν πρέπει να μπορεί να έχει μεγάλο το οικονομικό όφελο από την άρση των κυρώσεων. Έχει υποθεί και αυτό. Εδώ βρισκόμαστε. Αυτό ε, είναι ε, το παρόν. Θέλουμε να υπάρξει το νόμο δυνατόν κοινή επιτροπή. Στις 24 Ιανουαρίου τα είπε και ο πατός Και χθε. Μετά το Συμβούλιο είπα ότι κάνει πάντο δυνατόν ο πατός για την ε, διατήρηση της συμφωνίας ισχύ και την εξέβρεση μιας οικοδομητικής προσέγγισης. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Αρνάρ Μπαταμπάη, θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σας την άποψη για το μέλλον της ε, συμφωνίας με το Ιράν και τις πιθανές συνέπειες ε, για την ασφάλεια, την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια και άλλων υπήρων και φυσικά και την παγκόσμια ασφάλεια εν γέννη. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι τιμή που ξαναβρισκόμαι εδώ στις Βρυξέλλες. Μου ζητήσατε να μιλήσω λίγο για το πώς μπορούμε να αντιληφθούμε την προσέγγιση του Ιράν και τα όσα ωφέλει όσον αφορά τα πυρηνικά ζητήματα. Και είναι σαφές ότι όποτε τίθεται το θέμα, εμείς οι λεγόμενοι εμπειρογνώμονες ε, της ε, συμφωνίας, ε, πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη γιατί την αναφέρουμε, γιατί φαίνεται να κουράζει το θέμα. Ε, πρέπει να πω όμως ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να σταματήσουμε να το συζητούμε, διότι έχουμε ακόμα μια ευκαιρία να την ε, προφυλάξουμε και να την διατηρήσουμε ζωντανή και θα εξηγήσω και γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Προκειμένου να αντιληφθούμε λίγο καλύτερα την προσέγγιση του Ιράν όσον αφορά τα πυρηνικά ζητήματα και το πυρηνικό του πρόγραμμα, πρέπει να αντιληφθούμε και πρέπει να θυμόμαστε ότι η σημασία του προγράμματος αυτό για το Ιράν είναι ε, θέμα εθνικού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης. Και επειδή ακριβώ αυτό δεν ισχύει για τα πυρηνικά προγράμματα κάποιων ευρωπαϊκών χωρών, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι σημαντικό για το Ιράν. Κατά την άποψή μου έχει να κάνει με δύο σημαντικούς πυλώνες. Το ένα είναι η επιστημονική πρόοδος και το άλλο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα ως ένδειξη τεχνολογικής και επιστημονικής ε, ε, σύγχρονη αντιμετώπιση. Ε, μπορεί κανεί βέβαια να εντάξει πολλά επιχειρήματα για το κατά πόσον ισχύει, αλλά για του ηθήνοντε του Ιράν η επιστημονική πρόοδο είναι ε, υψή τη σημασία, ε, διότι ε, χώρα ε, η οποία θεωρεί ότι είναι περικυκλωμένη και συνεχώς ε, είναι έρμεο κυρώσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι νοοτροπία μπορεί να έχει. Και νομίζω ότι στο προηγούμενο πανέλ αναφέρθηκε ότι το πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ιατρικών ισοτόπων, άλλων καλλιτικών προϊόντων και το Ιράν όντως εκμεταλλεύεται την πυρηνική ενέργεια και για αυτές τις χρήσεις. Υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες επ' αυτού πριν από 17-18 χρόνια και από εκεί ξεκίνησε και το όλο θέμα για τη συζήτηση για τα πυρηνικά του Ιράν. Το Ιράν πάντα έλεγε ότι είναι στα πλαίσια της συμφωνίας μη διάδοσης η χρήση που κάνει και ε, είναι κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη εκτός Ιράν. Δεν το κρίνω αυτό, αλλά είναι γεγονός κατά την άποψή μου είναι το θρησκευτικό διάταγμα το οποίο ε, δημοσιεύθηκε από την υψηλότατη αρχή της χώρας, τον ε, Αγιατολά Χαμένη. Η παραγωγή, κατοχή και διάδοση ε, πυρηνικών όπλων μαζική ε, καταστροφή είναι κατά του Ισλαμικού νόμου. Αυτό δεν ε, ε, περνάει ω επιχείρημα στην Ευρώπη, δεν το πιστεύει κανεί, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε σοβαρή υπόψη. Νομίζω ότι αυτό που ήταν ένα κομβικό σημείο είναι ότι πριν από τη συμφωνία με το Ιράκ και την αρχή τη εφαρμογή τη υπήρχε η άποψη ότι δεν θα μπορέσει να κάνει πλουτισμό στο Ιράν το Ιράν. Και αυτή ήταν η μία προσέγγιση η οποία αποτέλεσε και το ένευσμα για την ιδέα αυτή για το κύρος, ε, για το ότι μας απαγορεύεται να κάνουμε το, αυτό το εγγυόμαστε στα μέλη της Συμφωνίας Μη Διάδοσης πυρονικών. Μέσα σε ένα-δύο χρόνια, το 2002-2003 και από εκεί και πέρα, το πυρηνικό ζήτημα ουσιαστικά έγινε ένα ζήτημα βάσει του οποίου οι δυτικέ οι παγκόσμιε δυνάμει ασκούν πιέσει προ το Ιράν και το Ιράν προσπαθεί να δείξει την ανθεκτικότητά του, να αντισταθεί και οι συζητήσει προφανώ πήγαν πολύ πέραν των πυρηνικών θεμάτων, διότι ανέκαθεν ήταν ε, το γεωπολιτικό ζήτημα στη Μέση Ανατολή το θέμα, αλλά το πυρηνικό ήταν το ένα θέμα μέσω του οποίου διοχετεύθηκαν όλα αυτά το χρησιμοποιήθηκαν για να επιβάλ, ε, χρησιμοποίησαν για να επιβάλλουν κυρώσεις ε, και να το περιορίσουν. Το Ιράν το εκμεταλλεύεται για να δείξει ότι αντιστέκεται, να προκαλέσει και να δείξει ότι ε, υπάρχει και ένας ανασταλτικός παράγων και φυσικά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το Ιράν παίζει με αυτή την έννοια της πυρηνικής απειλής. Πάντα λέει ότι δεν έχει ε, πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, το οποίο εγώ πιστεύω, αλλά πάντα υπάρχουν κάποιες αμφισημίες οι οποίες εν τέλει, όπως ε, σας είπα ήδη προηγουμένως, οδήγησαν και σε όλες αυτές τις συζητήσεις περί πυρηνικών. Και νομίζω το 2003 είχαμε τους τρεις ε, Υπουργών Εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου που πήγαν στην Τεχεράνη για να προλάβουν δύο πράγματα. Πυρηνική βόμβα από το Ιράν από την Ευρωπαϊκή Σκοπιά και την απειλή ε, μιας στρατιωτική κλιμάκωσης στην περιοχή. Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα αντίστοιχο σταυροδρόμι τώρα. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η προοπτική μιας ε, ε, επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ ή την αποχώρηση του Ιράν από τη συμφωνία και από τη συμφωνία μη διάδοσης και να επανέλθει στο θέμα της πυρηνικής απειλής. Και εδώ έχουμε μια διάσταση την οποία εκμεταλλεύεται πλέον το Ιράν για να πιέσει για τις, κατά των πιέσεων που του ασκούν. Και νομίζω ότι κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω όσον αφορά το πώς καταφέραμε να έχουμε τη συμφωνία με το Ιράν, σίγουρα το καθεστώς κυρώσεων που υπήρχε είχε οικονομικό αντίκτυπο, αλλά ο πολιτικός αντίκτυπος ο οποίος τελικά οδήγησε στην επίτευξη της συμφωνίας από πλευράς Ιράν ήταν ότι ε, θα εγκατέλειπαν την πολιτική μηδενικού εμπλωτισμού, το οποίο δέχθηκε ε, ο πρόεδρος Ομπάμα. Ε, αυτό λοιπόν ήταν αυτό που, το οποίο κατά την όποψή μου οδήγησε το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πόσα λεπτά έχω ακόμα, δύο, τρία, δύο. Ωραία. Πού βρισκόμαστε τώρα και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το Ιράν είναι σε κατάσταση πολιοργίας. Ξέρετε τι πιέσεις ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν και το Ιράν πιέζει σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι σε περιφερειακή διάσταση, κλιμακώνοντας κάποια πράγματα στον Περσικό κόλπο, απειλώντας ε, τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο δεύτερος πυλώνας είναι το πυρηνικό. Από τη μια πρέπει να τονίσω ότι αν το Ιράν πραγματικά ήθελε να φύγει από τη συμφωνία, Κατά την άποψή μου θα το είχε κάνει ήδη. Βλέπουμε λοιπόν ακόμα ότι υπάρχει διάθεση από πλευρά Ιράν να την προφυλάξουν τη συμφωνία παρά το γεγονό ότι υπήρξαν κάποια βήματα προ την άλλη κατεύθυνση. Κατά την άποψή μου, ε, οι επιθεωρητέ τη υπηρεσία ε, ατομική ενέργεια ακόμα δεν έχουν εκδιωχθεί από το Ιράν. Επομένω, όλοι ξέρουν τι κάνει το Ιράν. Το γεγονό ότι δεν του έχει διώξει είναι σαφή ένδειξη. Τώρα, κάποιε συστάσει. Πιστεύω ότι ο μηχανισμό επίλυση διαφορών έχει τον όρο επίλυση τη διαφοράς και επομένω είναι πολύ σημαντικό να επιληθεί το όλο θέμα. Όχι να αρχίσουμε να κατηγορούμε αλλήλου που θα είναι η διαφορά ή να το επεκτείνουμε απλώς για να συζητούμε που είναι ο μηχανισμός, αλλά να δώσουμε έμφαση στην επίλυση του θέματο. Και η επίλυση θα μπορούσε να προκύψει αν δώσουμε αντικίνητρα στο Ιράν για να μην πιέσει στην κλιμάκωση των υποχρεώσεων και ξέρω ότι έχει κουράσει και αυτό το θέμα, αλλά εδώ μόνο τιμωρίες μπορεί να έχουμε. Εάν δεν υπάρχουν κάποια αντικίνητρα για τις εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, δεν θα μπορέσει το Ιράν να λιώσει τα θέματα αυτά. Υπάρχουν θέματα περιφερειακής ασφάλειας, μπορεί να έχετε και τις ε, αμφιβολίες σας, αλλά εγώ θεωρώ ότι το Ιράν θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτά. Και τέλος, και πραγματικά τελειώνω, αναφερθήκαμε στις τρεις πρωτοβουλίες, ένα ευρωπαϊκό ε, μήνυμα θα ήταν να έχουμε τρει Ευρωπαίου ε, υπουργού Εξωτερικών μαζί με τον ύπατο εκπρόσωπο να πάνε στο Ιράν και να δείξουν ότι υπάρχει ένα ενωμένο ευρωπαϊκό μέτωπο κατά τη προσέγγιση των ΗΠΑ για τη συμφωνία με το Ιράν. Τουλάχιστον θα δώσει στο Ιράν μια ένδειξη ότι οι ε, Ευρωπαίοι τολμούν να κάνουν την πολιτική επένδυση στο θέμα αυτό. Συγγνώμη που μακρηγόρησα και φυσικά είμαι στη διάθεσή σα για περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μίξερ από τους σοσιαλιστές. Sorry. Thank you, Madam Chair. Uh, I have a couple of uh, questions. Uh, first... Μια-δυο ερωτήσεις. Ε, κάτι που συνδέεται με το προηγούμενο θέμα την παραμονή της υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν υπήρχαν προειδοποίησεις από διάφορες πλευρές ότι το Ιράν μήνες απήχε ε, από το να γίνει πλήρης ε, πυρηνική δύναμη. Και αμέσως μετά την συμφωνία, οι ίδιοι άρχισαν να παραπονιούνται για την βραχία χρονική διάρκεια της ε, συμφωνίας. Είπαν ότι καλή είναι προς το παρόν, αλλά τι γίνεται σε 10-15 χρόνια. Η ιδέα ήταν όμως ότι ακόμα και αν είχαμε καθυστέρηση της ε, πυρηνικής ας πούμε, πορείας του Ιράν για 10-15 χρόνια, θετικό θα ήταν. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν διαφορές. για το πώς μπορεί να επηρεάσει η κατάργηση της συμφωνίας την πυρηνική πορεία του Ιράν. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε λιγάκι. Τι διαφορές αντιλήψεις υπάρχουν μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής και Ρωσίας για το εγγύς μέλλον της συμφωνίας. Και τι σημαίνει αυτό το γεγονός ότι είχε βραχία διάρκεια η συμφωνία τι επιπτώσεις είχε στην, ε, στις στρατιωτικές δυνατότητες και πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν. Κάτι άλλο που συνδέεται με προηγούμενο σημείο. Κάποιος ομιλητής είπε ότι υπάρχουν διαφορές ε, στο πώς αξιολογούμε την απειλή που συνιστά το Ιράν σε ό,τι αφορά τη διάδοση των πυρηνικών. Η Αμερική σήμερα θεωρεί ότι βραχυπρόθεσμα δημιουργεί απειλή το Ιράν για τη μη διάδοση, ενώ η Ρωσία δεν συμφωνεί. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την διαφορετική προσέγγιση. Και ένας ομιλητής είπε ότι στην ε, δημόσια και πολιτική συζήτηση στην Ευρώπη εστιάζουμε κυρίως στην ανάγκη να διατηρήσουμε τη συμφωνία ως ε, μίζωνα πολιτική και διπλωματική νίκη, στην οποία συνεισέφερε τα μάλα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πως θα έπρεπε να εστιάσουμε περισσότερο στο μηχανισμό επαλήθευσης της ε, Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας και τι υποχρεώσεις του Ιράν ε, υπό τη συνθήκη μη διάδοσης, γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με, την, με τα πυρηνικά. Τι άποψη έχετε γι' αυτό. Merci pour les verts, Buchner. Κύριος Μπιούχνερ από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις εισαγωγικές πίσω παρεμβάσεις σας. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις ε, για την ανάπτυξη για τον πλούτο ακούσαμε πολλά. Κάτι ανησυχητικό και σημαντικό είναι ένα ερώτημα. Γιατί έχει τόσες ε, εσωτερικές δυσκολίες στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Η ελπίδα, ή να το πω αλλιώς, στο Ιράν ε, η Επανάσταση, το Συμβούλιο, το Επαναστατικό και για το Λάδες ε, έχουν πει ότι θα προχωρήσουν και το θέμα είναι να είναι καλύτερα τα πράγματα για το λαό λόγω της άρσης των κυρώσεων. Υπάρχει δηλαδή εμπιστοσύνη στη διεθνή κοινότητα προς αυτό. Έχουμε μετά τη δράση των ήπα. Ε, ε, ουσιαστικά έχει καυθεί λόγω των απειλών ε, των ΗΠΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν επαναεπιβληθεί πλέον οι κυρώσεις από την Αμερικανική πλευρά. Το θέμα είναι υπάρχει ε, πλειοψηφία που μπορεί να πιστεί στο Ιράν να ε, συνεχίσει να εμπιστεύεται την κοινότητα και αν ναι θα πρέπει να βρούμε τη δυνατότητα εμείς τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά να άρουμε τις κυρώσεις Το λέει και το έχει ξαναπεί πολλές φορές ε, και ο υπουργό ε, Εξωτερικών του Ιράν. Έχουμε αυτό τον ε, οικονομικό μηχανισμό, τον χρηματοδοτικό μηχανισμό που ουσιαστικά επιτρέπει πάρα πολύ περισμένες εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν πολύ ελάχιστο όγκος των συναλλαγών, αλλά είναι σημαντικό για τους Ιρανούς ως πηγή χρηματοδότης παρόλα αυτά. Αν θέλουμε λοιπόν κάτι να πετύχουμε, μπορούμε να μιλάμε για την πυρηνική τεχνολογία και να λέμε πολλά και είναι και η ειδικότητά μου και αν θέλετε ευχαριστώ να σας τα πω, αλλά από πολιτικές πλευράς δεν κάνουμε πολλά. Από πολιτικές πλευράς πρέπει να άρουμε τις κυρώσεις, αν θέλουμε κάτι να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Γουάλλας από την ΚΟΕ. Μία σύντομη ερώτηση και στους δύο μιλητές. Στο τελευταίο θέμα έθεσα, πριν μπείτε εσείς δηλαδή, έθεσα ένα ερώτημα στον κύριο Χίμπς, ας πούμε. Τον ρώτησα εάν η Ευρώπη είναι αβοήθητη. Αν δεν μπορεί να επιλύσει λόγω της Αμερικανής αντίθεσης τα προβλήματα με τη συνθήκη με το Ιράν ή αν μπορεί να κάνει περισσότερα. Ε, και απάντησε ότι ο μεγάλος φόβος για την Ευρώπη είναι οι κυρώσεις. Εσεί πιστεύετε ότι η Ευρώπη μπορεί να πει στου δύο παίχτε, Κοιτάξτε. Η αμερικανική θέση δεν είναι προς το συμφέρον της ειρήνης, δεν είναι αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι. Πιστεύετε ότι θα έχει το θάρρος η Ευρώπη να πάρει μια ανεξάρτητη θέση ως προς Αμερικανούς. Να κάνει το σωστό για να μπορέσει να επανέλθει η συμφωνία και να διασωθεί η συμφωνία, να διασώσουμε τη συμφωνία. Ο κύριος Αουστροβίσιους από το Renew Europe. Ευχαριστώ. Εγώ έχω την αντίθετη άποψη. Μερικές φορές οι οικονομικές κυρώσεις είναι αναπόφευκτες. Πρέπει να επιβληθούν για να σταματήσουμε τις κακές συμπεριφορές χωρών που είναι υπέρ της διάδοσης και του εμπλουτισμού του ουρανίου. Που είναι ένα βήμα πριν αναπτύξουν πυρηνικά όπλα που είναι τεράστια περιφερειακή απειλή, για να μην πω και παγκόσμια απειλή. Σε ποιο βαθμό λοιπόν η πολιτική με τις οικονομικές κυρώσεις μπορεί να εμποδίσει το Ιράν από το να προχωρήσει, να περάσει στον εμπλουτισμό και να διαδώσει τα πυρηνικά. Ε, μπορεί να, οι κυρώσεις να τους σταματήσουν γιατί δεν, δεν θα έχουν τους οικονομικούς πόρους για να προχωρήσουν με το πρόγραμμά τους. Επίσης το Ιράν είναι πιο προχωρημένο στην ανάπτυξη πυράβλων. Το έχουν πει πολλέ περιφερειακές, πολλέ χώρε της ε, περιφέρειας και θεωρείται όλο και μεγαλύτερη απειλή. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ε, πυράβλων δημιουργεί πρόβλημα. Το Ιράν δίνει πυράβλους σε ορισμένε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως ε, η Χεσμολά, οι οποίες επιτίθενται στο Ισραήλ. Αυτά τα πυραυλικά συστήματα είναι αρκετά προχωρημένα. Αρκετά προηγμένα τεχνολογικά και γίνονται και μεγαλύτερες προσπάθειες περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των συστημάτων για τα επόμενα χρόνια. Αυτό τι σχέση έχει με την ε, συμφωνία, δεδομένου ότι το Ιράν προχωράει ή θέλει να προχωρήσει στο πρόγραμμα εμπλουτισμού του ουρανίου. Δεδομένης αυτής της ε, βούλησης ε, πρέπει να ανησυχήσουμε για τους πυράβλους του Ιράν. Από το ΕΛΚ, ο κύριος Πέτερς. Ευχαριστώ τους ομιλητές για τις πληροφορίες ε, που είναι πολύ σημαντικές. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ διαβάζω πάντα όλα τα έγγραφα που εγκρίνουμε και εγκρίθηκε ένα έγγραφο για την εφαρμογή της, για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας. Στο σημείο 56 λέμε κάτι. Αυτό που συμφωνήσαμε στο Στρασβούργο. Θα πρέπει, είπα, η εκπρόσωπος να χρησιμοποιήσει όλη την πολιτική και διπλωματική δυνατότητα που έχει, ούτω ώστε να διατηρηθεί η συμφωνία και να υπάρξει στρατηγική μείωση των πυρηνικών. Και θα πρέπει η Ευρώπη να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητά τη που έχει διπλωματικά, ούτω ώστε να συνομιλήσει με όλου του εταίρου και έχει αυτή τη δυνατότητα που θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσει πλήρω, 100%. Αυτό συμφωνήσαμε στο σημείο 56 του κειμένου. Είπατε ήδη ότι η δράση της είπα της εκπροσώπου ή του είπα του εκπροσώπου απέναντι στις άλλες χώρες είναι κάτι που το έχουμε ζητήσει και εμείς. Το θέμα είναι, αρκεί αυτό. Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα για να βρούμε λύση. Το μόνος τρόπος για να βρεθεί λύση. Ή πρέπει να γίνει και κάτι παραπάνω. Κυρώσεις δηλαδή. Χρειάζονται κυρώσεις ή αυτό που συμφωνήσαμε στο Στρασβούργο αρκεί. Αρκεί ή όχι. Θα δώσω το λόγο στους παρεμβαίνοντες. Άκουσα και εγώ σήμερα το πρωί πολλά πράγματα, διάφορους ισχυρισμούς ότι το Ιράν θέλει, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα κανονικό κράτος και δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις, ή Το θέλει κάτι τέτοιο το Ιράν. Όταν θέλει να εξάγει την ε, επανάστασή του, υποστηρίζοντας και τρομοκρατικές ομάδες και υποσκάβοντας τη σταθερότητα της ε, περιοχής. Υπάρχει αντίφαση, αυτή η ένταση. Επίσης, θα ήθελα να μου απαντήσουν οι συμμετέχοντες στο πάνελ την άποψή τους για αυτά τα θέματα, καθώς και για τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με μια γενική παρατήρηση καταρχάς και μετά να περάσω σε πιο συγκεκριμένε απαντήσεις. Καταρχάς, γιατί η συμφωνία με το Ιράν και πού επικεντρώθηκε. Αυτή είναι μια πυρηνική συμφωνία με ένα σκέλος με Δεν ήταν μια συμφωνία η οποία σχεδιάστηκε για την περιφερειακή σταθερότητα τότε ε, η απόφαση αφορούσε και κατά πόσο ήταν εφικτή και πώς μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία η οποία είναι πολύ εύρωστη. Αν τη δείτε με όλα τα παραρτήματα και τις λεπτομέρειές της, είναι πάρα πολύ διεξοδική όπως σας είπα στην αρχή, δίνει πρόσβαση για επαλήθευση και ίσως εδώ και σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν και για τη φάτουα αυτό το διάταγμα το ε, Ισλαμικό, ε, ε δεν θέλουν να έχουν βόμβα, και υπήρχε και εμπιστοσύνη για επαλήθευση, το σημειώσαμε, είδαμε όμως και κάποιες δραστηριότητες και υπάρχει ένα πάρα πολύ ε, ισχυρό καθεστώς επαλήθευσης ε, βάσει του οποίου υποβάλλει εκθέσεις η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες της συμφωνίας επίσης ε, βάσει αυτού δέχτηκαν να άρουν τις κυρώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πω ότι το έχει κάνει από πλευρά της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άρει τις ε, κυρώσεις της βάσει της συμφωνίας. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία επίσης συλλάβουν με τη συμφωνία, αλλά δεν έχουν εισαχθεί νέες καθόλου κυρώσεις. Αυτό που συλλεύει είναι ότι ένας από τους συμμετέχοντες της συμφωνίας αποφάσισε για πολιτικούς λόγους μετά τις εκλογές να αποσύρει τη συμμετοχή του στη συμφωνία. Μια συμφωνία την οποία, όπως ανέφερα, ε, θεωρούμε ότι είναι λυπηρή και εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι είναι λυπηρή, διότι θεωρούσαμε ότι με αυτή τη συμφωνία, με όλους τους συμμετέχοντες ε, να δέχονται τα θέματα, η περιφέρεια θα ήταν πιο ασφαλής. Αυτό που σημαίνει επίσης ότι ε, ξαναέχουμε κυρώσει από τις ΗΠΑ και ε, εξοεδαφικές συνέπειες αυτών των κυρώσεων. Εμείς είραμε τις κυρώσεις μας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε στις επιχειρήσεις μας τι θα κάνουν. Δεν είμαστε ε, κρατική οικονομία και εάν ε, οι επιχειρήσεις κάνουν υπολογισμούς για κίνδυνο και εκτίθενται σε αμερικανικές αγορές και είναι και έρμεους εκκυρώσεις από τις αμερικανικές αρχές, αυτό σημαίνει ότι θα λάβουν κάποιες αποφάσεις. Αυτό είχε κάποιο αντίκτυπο, το γνωρίζουμε και προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με πιθανά ωφέλη ε, για άρση κυρώσεων με τους Ιρανούς εταίρους. Ε, ο ύπατος εκπρέσεως αναγνώρισε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει άρση κυρώσεων για το Ιράν, αλλά όσον αφορά τις υποχρεώσεις του το, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Τώρα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορεί να κάνει το Συμβούλιο, να αλλάξει η νομοθεσία και να άρει τις κυρώσεις και όχι να υποχρεώνει τον κόσμο να έχει εμπορικές σχέσεις ή όχι. Αναφέρθηκε και ω ε, μια σημαντική οδό η συμφωνία για λαεθαρρύνη αυτή τη μορφή στο εμπόριο, γιατί είναι και ένα σχέδιο για οικονομικέ ανταλλαγές, το οποίο προστατεύεται από πιθανέ εξοεδαφικές κυρώσει. Και υπάρχουν συζητήσει για το πώ μπορούμε να τα αναβαθμίσουμε τα πράγματα, πώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα, κυρίως όσον αφορά το ανθρωπιστικό εμπόριο, αλλά εν τέλει όχι απαραίτητο και μόνο γι' αυτό. Όσον αφορά τώρα τις ε, συνέπειες της συμφωνίας ε, και τον κίνδυνο ε, για διάδοση πυρονικών, όταν συνάφθηκε η συμφωνία το 2015, είχαμε εκτιμήσει ότι θα είχαμε ένα διάστημα δύο μηνών, που είναι σύντομο διάστημα για να ξεκινήσουν τα πάντα. Το Ιράν είχε εφαρμόσει τις υποχρεώσεις του για τρία χρόνια και είχαμε περάσει λοιπόν το ε, διάστημα του ενός έτους ε, για τον κίνδυνο να μην τηρήσει τη συμφωνία Μειώθηκε όμως το διάστημα στο οποίο θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα με τη συμφωνία, αλλά και πάλι εκτιμάται στον ένα χρόνο γιατί έχει να κάνει και με τεχνικό εξοπλισμό, θα πρέπει να αναπτυχθεί τεχνικός εξοπλισμός και ακόμα βρισκόμαστε λοιπόν περίπου στον ένα χρόνο από τη στιγμή που αποφασίσει να μη, να συμμετέχει. Όσον αφορά βαλιστικού πυράβλους, ένα θέμα το οποίο ετέθη, έχει συζητηθεί και σε ψήφισμα το Λομπέλο Λεθλό τη Συμβουλία Ασφαλεία για τα πυρηνικά όπλα. Η δική μας η θέση και πάλι είναι ότι με πλήρη εφαρμογή της συμφωνία με όλου του συμμετέχοντες ο κίνδυνο θα μειωθεί για τους πυράβλου. Διότι όταν δεν υπάρχει συσκευή πυρηνική για να ε, ε, εξοπλίσει κάποιο με βαλιστικό πύραυλο δεν θα υπάρχει πύραυλος. Αυτά είναι και τα επιχειρήματα και οι λόγοι για τους οποίους λέμε ότι έχει υπάρξει συμπόρφωση αυτά τα τρία χρόνια από πλευρά Ιράν και είχε αποτέλεσμα η συμφωνία, βοήθησε και συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα. Τώρα βέβαια είναι πιο σύνθετα τα πράγματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και εδώ ερχόμαστε στις προσπάθειες του είπα του εκπροσώπου, νομίζω στις αρχές του έτους όταν ε, είδαμε και πόσο ευαίσθητο και ανησυχητικό είναι το πρόβλημα και μπορεί να υπάρξει περιφερειακή κλιμάκωση μετά από τη δολοφονία του Σουλεμάνη και τις επιθέσεις με επιράβλους που έγιναν ε, αμέσως ε, συνεκλήθη έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Ο ύπατος εκπρόσωπος πήρε και εντολή να πάει στην περιοχή να συζητήσει με τους εταίρους ε, ε, τα θέματα της περιφερειακής ασφάλειας μέσω μέτρων δημιουργίας εμπιστοσύνης, μέσω συγκεκριμένων βημάτων που θα βοηθήσουν στο διάλογο και το ταξίδι του στην Τεχεράνη ήταν τμήμα αυτή τη ευρύτερη ε, ε, αποστολή. Μίλησε φυσικά και για τη συμφωνία, αλλά ήταν τμήμα τη ευρύτερη αποστολή του και συνεχίζει να παρακολουθεί το ζήτημα. Όσον αφορά τη συμφωνία με το Ιράν, μετά που ξεκίνησε το DRM από τους ε, τρεις της ευρωπαϊκή Ένωσης, όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, αυτοί θέλουν να διατηρήσουν την τη συμφωνία και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο. Από τη μια έχουμε σοβαρή ανησυχία που έθεσαν οι, οι τρεις για του πυρηνικά ζητήματα, αλλά θέλουμε να δούμε και κατά πόσο μπορούν να γίνουν κάποιες κινήσεις και σε οικονομικό πλαίσιο. Κάτι το οποίο θα δώσει και κίνητρα στο Ιράν και να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Να δω λίγο αν έχω απαντήσει σε όλα, αλλά νομίζω ότι απάντησα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το τελευταίο λεπτό που μας έμεινε, τα παταμπάει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Για τον κύριο Μίξερ. Τα είπατε πολύ ξεκάθαρα ότι αρχικά υπήρχε ο κίνδυνος ε, της διάλυσης ε, και θέλω να σας πω ότι αν λυθεί το ζήτημα με τα λεγόμενα sunset της ρήτρη σταδιακής κατάργησης όλα θα είναι καλύτερα. Σε ό,τι αφορά αυτές τις ρήτρε sunset ε, έχουμε τον Ιρανό προεξωτερικό που έχει πει αυτά που είπε που δεν θα τα δεν είχε τη στήριξη των αρχών της χώρας που λέει ότι θα τεθεί ε, υπόψη του Κοινοβουλίου το πρόστο πρωτόκολλο για την επικύρωσή του, όχι το 2023 αλλά νωρίτερα. Όλα αυτά ε, μπορούν να ε, ληφθούν υπόψη λοιπόν. Και υπ' αυτήν την έννοια απειλή να γίνει πυρηνικό κράτος στο Ιράν μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ απλά. Αρκεί κανείς να ακούει προσεκτικά αυτά που προσφέρει το Ιράν. Βέβαια σε αντάλλαγμα ε, της άρσης των, ε, με αντάγμα την άρση των κυρώσεων. Επομένως, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπει σε ένα νέο πλαίσιο ε, το όλο πράγμα για να έχουμε επιτυχία. Πρέπει απλά να μείνουμε στις τεχνικές πτυχές. Ο κύριος Μπίχνερ μίλησε για την εσωτερική διάσταση στη χώρα. Πρέπει να σας πω ότι η τη επανάσταση και η διοίκησή τους ουσιαστικά δεν είναι κατά της, ε, του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου. Υπήρξε απλά ένας ανταγωνισμός ε, ποιος θα είναι ο βασικός δικαιούχος, ποιος θα είναι ο αποδέκτης αυτής της οικονομικής άνθησης ε, που περιμέναμε θα, είχε, ε, που θα γινόταν για τη χώρα. Αυτό ήταν το θέμα. Ήταν θέμα σχετισμού δυνάμεων, καμία σχέση με το αν ήταν υπέρ ή κατά. Ε, και κάτι άλλο που είπατε, ότι πρέπει να δοθούν επιχειρήματα, ε, ώστε να μπορούν αυτοί που είναι υπέρμαχοι του κοινού οργανωμένου σχεδίου να δίνουν αυτά τα επιχειρήματα και να πείθουν τον κόσμο ότι ναι, είναι κάτι καλό. Ο κύριος Γόλης, μιλήσατε για αλλαγή παραδείγματος. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, για να αναπτύξει τη στρατηγική της αυτονομία σε τέτοιου είδους παγκόσμια ζητήματα. Αλλά γι' αυτό θα χρειαστεί μια ακόμη γενιά, θα έλεγα, πολιτικών ελίτ. Εμείς ε, βλέπουμε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον για το διατλαντικό σχεδεσμό και όταν ε, τα πράγματα κάπως ε, βγαίνουν ίσως από κάποια πλαίσια και προκύπτουν κάποιες εντάσεις, όλοι επανεπιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους ε, σε αυτό το δεσμό. Το θέμα βέβαια είναι η μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Υπάρχει πίεση από πλευρά Αμερικανών στου Ευρωπαίου και δυστυχώ ε, επιτυχημένη πίεση. Πώ θα γίνει λοιπόν αυτή η αλλαγή, παραδείγματο δεν ξέρω. Μάλλον πρέπει να έρθει η επόμενη γενιά πολιτικών στην Ευρώπη. Και τα τελευταία δύο σημεία του κ. Στρεβίσιο καταρχά. Οι κυρώσει ως μέσο αλλαγής συμπεριφορών. Πράγματι, υπήρξαν κράτη που άλλαξε η συμπεριφορά τους ε, όταν ήταν ε, σε ισχύ το καθεστώ ε, επιβολή και δεν άλλαξε όμω το Ιράν πολιτική, άλλαξαν Ευρωπαίοι πολιτικοί ε, απέναντι στο Ιράν, όπως και το ίδιο έκαναν άλλα κράτη απέναντι στο Ιράν. Και ο σχεδιασμός είναι αυτός των κυρώσεων. Δεν αλλάζει η χώρα. Είναι πώς οι άλλοι συναλλάσσονται με αυτή τη χώρα. Και γι' αυτό θεωρώ ε, ότι έτσι αιτιολογείται το ότι γιατί δεν βλέπουμε κάποια θετική ε, στάση και ανταπόκριση απέναντι στις κυρώσεις αυτές των Αμερικάνων. Η επίσκεψη του είπα του εκπροσώπου αναρκεί, ναι. Ακούστε, είμαστε σε ένα σημείο που χρειάζεται οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνη. Μακάρι να μην ήταν έτσι. Μακάρι να το είχαμε ξεπεράσει, όπω πριν κάποια χρόνια. Όμω τώρα χρειάζεται το Ιράν να δει ένα μήνυμα, ένα δείγμα ότι έστω η Ευρώπη είναι ενωμένη. Ή τέλο πάντων η βασική υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων για αυτό το σχέδιο. Άρα οι ευρωπαϊκέ τρίτε χώρε, οι τρει ευρωπαϊκέ χώρε και ο του πρόσωπο ε, χρειάζεται η Ένωση. Δεν το λέω ότι είμαι στι Βρυξέλλε. Χρειάζεται αυτή την όθηση Ένωση Και ο ύπατος εκπρόσωπο και τώρα και η ύπατη εκπρόσωπος τα τελευταία δύο χρόνια ήταν το μόνο πρόσωπο το οποίο αντιστάθηκε στις πιέσει των Αμερικών Δεν άκουσα να λένε τίποτα οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, όπως το έκανε η Φρεντερίκα Μογκερίνη και τώρα ο Ζωζέ Μπορέλ. Αυτό νομίζω είναι ο δρόμος ε, προ τα... Ε, χρειάζεται όμω τα τρία ευρωπαϊκά κράτη να υποστηρίξουν, να βάλουν πλάτη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό και μετά από κάνα δύο λεπτά να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερισχές διάταξης για την Κορετική Χερσόνησο. Genau, also allerdings, ich habe, glaube ich, nur deine, oh, doch, die E-Mail habe ich ja auch. Aber dann, ich melde mich nochmal wegen... Super, wenn du da bist und ich bin sehr interessiert dran, was du so... Nee, natürlich, das, was da los ist.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 μας. Euh, euh, Περνάμε στο σημείο που αφορά την ανταλλαγή απόψεων για την ασφάλεια στην Ανατολική Ασία και τις προοπτικές αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου. Καλωσορίζω τους ομιλητές μας, τον κύριο Ραμόν Πατσέντο, Πατσέκο Πάρδο, πρόεδρο της ε, KFVUB, του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών, και τον κύριο Ράινχολντ ε, Μπρέντερ, ε, επικεφαλής ε, Ιαπωνίας, Κορέας, Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και Ειρηνικού στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας. Ε, Εξωτερική δράση, συγγνώμη. Οι παράνομε πυρηνικέ δραστηριότητε τη Βόρεια Κορέα είναι πηγή ανησυχία για τη διεθνή κοινότητα. Μετά την αποχώρησή τη το 2003 από τη συνθήκη μη διάδοση, <clears throat> επιτάχυνε το πρόγραμμα πυρηνικών και μόνο τρία χρόνια μετά, το 2006, έκανε το πρώτο, την πρώτη πυρηνική δοκιμή. Την επόμενη δεκαετία έκανε πέντε πυρηνικέ δοκιμέ. Ε, εν συνεχεία, το Συμβούλιο Ασφαλεία ε, κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα και τα πυρηνικά προγράμματα ε, και να σταματήσει τι συναφεί δραστηριότητε. Οι κυρώσει συνοδεύουν αυτά τα ψηφίσματα και θέλουν να εμποδίσουν τη Βόρεια Κορέα να αναπτύξει περαιτέρω την πυρηνική τεχνολογία και το πρόγραμμα πυράβλων. Πολλέ χώρε, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επέβαλαν κυρώσει αυτόνομε ε, για να αυξηθεί η πίεση στη Βόρεια Κορέα, ούτω ώστε να συμμορφωθεί με τι διεθνεί υποχρεώσει τη. Ο πρόεδρο τη Νότια Κορέα ε, υποστηρίζει τι διεθνεί κυρώσει εναντίον τη Βόρεια Κορέα, έχει μία όμω πιο συμφιλιωτική προσέγγιση και έκανε σημαντικέ προσπάθειε για να βελτιώσει τι σχέσει μεταξύ των δύο χωρών, Βόρεια και Νότια Κορέα. Η πρώτη ε, Σύνος κορυφής μεταξύ Αμερικής και Βόρειας Κορέας έγινε το 2018 και οδήγησε σε μια κοινή δήλωση που υπογράφηκε στη Σιγκαπούρη, ε, ούτω ώστε η Βόρεια Κορέα να κάνει μια προσπάθεια αποπυρικοποίηση ε, τη Βόρειας, της χερσονήσου της Βόρειας της, Κορέας. Δυστυχώς, ε, οι προσπάθειες για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις είπα, Βόρειας Κορέας ε, ατύχησαν. Μετά την αποτυχία της συνεδρίας της Στοκχόλμης, ε, φαίνεται ότι η Βόρεια Κορέα δεν είναι έτοιμη να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά είναι ανοιχτή η πόρτα για μελλοντικέ διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Μερικές... Ε, όμως όλα αυτά εξαρτώνται από τις αμερικανικές αποφάσεις. Ε, οι Αμερικανοί είναι στραμμένοι προς την Ασία και τον ειρηνικό, τον ε, ειρηνικό για τους ε, πυράβλους και στην περίπτωση που οι Αμερικανοί αποφασίσουν στην στο ε, να αναπτύξουν νέους βαλιστικούς ε, πυράβλους ε, που θα έχουν εμβέλεια 1.800 με 2.400 χιλιόμετρα. Αυτό ε, θα, τους, θα καθιστούσε την πιόν ε, πιο προσπελάσιμη και επομένως οποιαδήποτε διπλωματική λύση απομακρύνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντωμεταξύ δεν έχει στρατιωτική παρουσία ούτε σύστημα συμμαχίας στην Ανατολική Ασία ε, σε περίπτωση που διαπραγματεύσεις ε, ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας φτάσουν σε νέες ε, συμφωνίες, τότε η διάλυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας θα ήταν τεράστιο, μια τεράστια πρόκληση οικονομική και τεχνική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτό μπορεί να κάνει είναι να χρηματοδοτήσει τη διαδικασία πυρηνικοποίηση ε, σε περίπτωση που συμφωνήσουν ΗΠΑ και Βόρεια Κορέα και θα μπορούσε να παράσχει επιθεωρητές για να διαπιστώσουν κατά πόσο διαλύεται το πυρηνικό οπλοστάσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει μια ιδιαίτερη θέση, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική της ε, πραγματογνωμοσύνη και να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας και άλλων μερών που ενδιαφέρονται άμεσα από την ε, συμφωνία αυτή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πατσέκο Πάρτο για να μας πει την άποψή του για τις προοπτικές για την ένταξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας και για πιθανή συμφωνία με σκοπό την αποπυρηνικοποίηση της χερσονήσου της Κορέας. Και συνεχεία θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπρέντερ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση ε, ποιες είναι οι προοπτικές αποπυρηνικοποίησης της α, Χερσονήσου, της Κορέας και της Βόρειας, και της Βόρειας Κορέας. Ε, ε, start by talking... Θα ήθελα Εδώ Να σας εξηγήσω γιατί η Βόρεια Κορέα, η Βόρεια Κορέα έχει ένα πρόγραμμα πυρηνικών, κάτι που απειλεί το καθεστώς της συνθήκη μη διάδοσης και ποιο είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μπορούμε να παίξουμε κάποιο ρόλο για να πείσουμε την Βόρεια Κορέα να οδηγηθεί στην αποπυρηνικοποίηση. Ε, το πρόγραμμα το πυρηνικό τη Βορείας Κορέας δεν είναι καινούριο. Ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 60. Το 2003 η Βόρειος Κορέα έφυγε από τη συνθήκη μη διάδοση και τότε έγινε επιτάχυνση των εξελίξεων για ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματο. Ε, μιλάμε για 20 χρόνια προγράμματο εμπλουτισμού του ουρανίου. Να σας πω αν πιστεύω ότι είναι πιθανή όχι από πυρηνικοποίηση. Ακόμα και ένα βήμα προς την αποπυρηνικοποίηση είναι μια μακρόπνοη διαδικασία και δεν θα απασχολήσει μόνο μια Αμερικανική κυβέρνηση. Θα απασχολήσει και την ε, Νότιο και τη Βόρειο Κορέα. Και την Νότιο Κορέα, συγγνώμη. Καταρχάς, ε, γιατί αναπτύσσει πυρηνικό πρόγραμμα για λόγους αποτροπής. Το είδαμε και στην Μέση Ανατολή, που δεν είχαν πρόγραμμα πυρηνικών. Ε, πρόσφατα ασχολούνται με κάτι τέτοιο. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ε, η στρατιωτική παρουσία ε, των Αμερικανών, η στρατιωτική ισχύ τη Νότια Κορέας, το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας ε, γίνεται και για λόγους αποτροπής. Και για να μην επιτρέψει στους Αμερικανούς να σκοτώσει τα ηγετικά στελέχη του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας Επίση, υπάρχει ένα θέμα νομιμότητα που απορρέει από αυτό το πρόγραμμα, σε, αυτή την, σε αυτόν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στι δύο Κορέε. Η Νότιο Κορέα είναι μεγάλη οικονομική δύναμη, ε, η ήπια δύναμη. Ε, και η Βόρειο Κορέα τι έχει, πυρηνικά όπλα για να αναγνωριστεί ο σημαντικός παίχτη στην περιοχή. Ε, γιατί, κοιτάξτε, αν δεν είχε αυτή η χώρα τέτοια πυρηνικά, δεν θα κάναμε τόσε συζητήσει ε, για τη Βόρεια Κορέα. Ούτε εμεί, ούτε οι Αμερικανοί. Υπάρχει και το θέμα τη εξέβρεση πόρων, ε, χρήματο. Ε, όσοι έχουν ε, πυρηνική τεχνολογία ε, την εξάγουν και η Βόρεια Κορέα την εξάγει κυρίω στη Μέση Ανατολή και εξάγει και όπλα μαζική καταστροφή. Αλλιώ θα ήταν πολύ πιο δύσκολο ε, για το καθεστώ να επιβιώσει χωρί αυτή τη δραστηριότητα από την οποία εισπράττει βέβαια. Επίσης, ε, αυτό συνδέεται με τον ιδρυτή της ε, δυναστείας, τον παππού και τον πατέρα του τρέχοντος ε, ηγέτη του Κιμ. και ο σημερινός ηγέτης θέλει να συνεχίσει την κληρονομιά του παππού και πατέρα. υπάρχει λοιπόν και οικογενειακή αυτή παράδοση. Γιατί ε, η Βόρειο Κορέα είναι μεγάλη απειλή για το καθεστώς της ε, Συμφωνία Μη Καταρχά, Καταρχάς, ε, γιατί διαδίδει πυρηνικά επί δεκαετίε κυρίω στην Μέση Ανατολή. Επίσης, εξάγει πραγματογνωμοσύνη στο Ιράν, Φερρυπίν. Αναφέρθηκε στο προηγούμενο τμήμα, στην Συρία, το, στην Αίγυπτο, το παρελθόν, στη Λιβύη, σε πολλέ χώρε στον κόσμο εξάγει αυτή την γνώση, την πραγματογνωμοσύνη. Έχουν φιλοξενήσει χώρε αυτέ πυρηνικού επιστήμονε από τη Βόρεια Κορέα. Ε, για να τους βοηθήσουν να χτίσουν πυρηνικές εγκαταστάσεις. Επίσης, η Βόρειος ε, Κορέα έφυγε από το NPT το 2003 και αυτό είχε σημαντικές ε, συνέπειες και διπλωματικά. Είναι κράτος παρείας, αποδιοπομπαίο κράτος η Βόρειος Κορέα, έχει κυρώσεις, παρόλα αυτά επιβιώνει. Ε, και μάλιστα οικονομικά είναι σε καλύτερη θέση και πολιτικά ε, είναι σε καλύτερη θέση από όταν το 2003. Επίσης, ε, θέτει και το παράδειγμα σε άλλες χώρες που... και εμπνέει άλλες χώρες που θέλουν να φτιάξουν πυρηνικά. Γιατί αν λένε άλλες χώρες, ας πούμε, αφού μπορεί να το κάνει η Βόρειος Κορέα, μπορεί να το κάνω κι εγώ. Άρα είναι ένα αρνητικό παράδειγμα, κατά τους Ευρωπαίους βέβαια. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να κάνει. Αυτή τη στιγμή ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις και όταν υπογραφεί η συμφωνία είτε με τον Τραμπ είτε με οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση είτε μέσα στο 2020 σε πέντε χρόνια. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να και τα κρατημέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν τη συνθήκη με διάδοση. Η Βόρειο ε, Κορέα, είτε σα φαίνεται πιστευτό ή όχι, το λαμβάνει υπόψη αυτό. Ε, ακόμα και αν έχει φύγει, το γεγονός ότι συζητιέται το κατά πόσον σέβεται τη συμφωνία ε, την ενδιαφέρει. Επίσης, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να στραφούν διπλωματικά, να τίνουν χείρα διπλωματική προς την ε, Βόρεια Κορέα. Ο πολιτικός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βόρειος Κορέα, Βορείου Κορέας δεν έχει λειτουργεί, δεν υπάρχει. Κακό κατά τη γνώμη μου, γιατί λειτουργεί καλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πει στη Βόρεια Κορέα γιατί θα πρέπει να πάει προ την αποπυρηνικοποίηση, γιατί την ενδιαφέρει την Ευρώπη, γιατί την ενδιαφέρει το γεγονό ότι υπάρχει διάδοση ε, προ τη Μέση Ανατολή. Δεν χρειάζεται να στρέφεται μόνο προ την Νότιο, Νότιο Κορέα ή την Αμερική ή Ευρώπη. Μπορεί να απευθυνθεί κατευθείαν στη Βόρεια Κορέα. Επίσης, ε, και μπορεί να στραφεί και σε άλλες οργανώσεις. Ε, υπάρχουν και άλλες ε, οργανώσεις, ΜΚΟ και τα λοιπά, που τις ενδιαφέρει και η μη διάδοση και μπορεί να τη στηρίξει οικονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουν την αποπυρηνικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κατευθύνει τη χώρα αυτή προς την αποπυρηνικοποίηση. Δεν πρέπει να το κάνει από μόνη της. Θα χρειαστεί πίεση και πολλές χώρες και φορείς οι οποίοι θα την πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ε, διπλωματικής οδού όπως γίνεται σήμερα. Παρότι τους τελευταίους μήνες η διπλωματία ε, έχει σοπάσει, μετά τις εκλογές που θα έχουμε μέσα στο 2020 αργό, ε, φέτος ε, στην Αμερική, η διπλωματία θα ενισχυθεί Επίσης, ο ηγέτης της Νότιου, της Νοτιού Κορέας έχει ακόμα δύο χρόνια μπροστά του και στηρίζει αυτή τη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή μιας συμφωνίας, η οποία τελικά θα επιτευχθεί μεταξύ Βορείου Κορέας και ΙΠΑ, αυτή η συμφωνία θα έχει δέσμευση της Βόρειας Κορέας να αποπυρηνικοποιηθεί και θα έχει τη λέξη αποπυρηνικοποίηση. Η Γαλλία, ας πούμε, ε, επίσης, έχει τέτοια στάση προώθηση πυρηνικοποίηση. Η Γαλλία θέλει να βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα να διαλύσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς επιθεώρησης υπό την αιγίδα της ε, ατομικής υπηρεσίας, συγγνώμη, από τις την της ε, Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας και θα πρέπει τα κράτη-μέλη και οι διεθνεί οργανώσει να εμπλακούν και να στείλουν τους επιθεωρητές του επιτόπου στη Βόρεια Κορέα. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε πακέτο κινήτρων με βοήθεια, οικονομική βοήθεια, ενεργειακή ενδεχομένω βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κληθεί να πει την άποψή τη ε, για το σχεδιασμό του πακέτου, καλό θα ήταν να πει πώς πρέπει να διαμορφωθεί αυτό το πακέτο. Επίσης, η, Ρωτία, η Βόρειος Κορέα σε περίπτωση που πάει προς την κατάργηση των πυρηνικών όπλων θα ζητήσει να κρατήσει τα πυρηνικά της για ειρηνικούς σκοπούς. Τι θα γίνει με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να υπάρξει μια μετάβαση ε, αυτών των εγκαταστάσεων από τη σημερινή τους χρήση σε μια μελλοντική χρήση για ειρηνικούς σκοπούς. Ε, και εκεί θα πρέπει να μπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μπορούμε να πετύχουμε τώρα την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας. Στο εγγύς μέλλον όχι είναι η απάντηση σε δύο-πέντε χρόνια. Αλλά αν υπάρχει συμφωνία με τους Αμερικανούς, η οποία είναι ρεαλιστική, και θα μιλήσουμε περισσότερο παρακάτω για αυτό το θέμα, η συμφωνία θα έχει και μια δέσμευση της Βόρειας Κορέας προς την αποπυρηνικοποίηση. Ε, θα δεσμευτεί λοιπόν προς αυτό η Βόρειος Κορέα και ως ενδιάμεση θέση θα πρέπει να υπάρξει η παναχώρηση ε, του πυρηνικού προγράμματος ε, της ε, Βόρειας Κορέας. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει η αποπυρηνικοποίηση βαθμιδών. Καθ... Είναι πολύ πιθανό να γίνει λοιπόν αυτή η διαδικασία, εφόσον υπογραφεί η συμφωνία, βαθμιδών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρέντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σας παρουσιάσω και την προεπτική τη Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επί του θέματο. Όπως γνωρίζετε, η Παγκόσμια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωση του 2016 αναγνωρίζει ότι στον σύνθετο και ολοένα και πιο περίπλοκο κόσμο χρησιμοποιούνται ε, όπλα και για το καλό και για το κακό. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει για τη σταθερότητα στην ε, Ασία. Το 40% του εμπορίου ε, περνάει από την ε, νότια Κινέζικη θάλασσα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και εκεί επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας σήμερα. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την προσέγγιση των ΗΠΑ για το πυρηνικό ζήτημα Κάποια τα έχουμε τονίσει. Η ουσία είναι ότι όσον αφορά την πολιτική μας ε, για την ε, Βόρεια Κορέα, ε, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια στάση ως, που, την οποία περιγράφουμε ως κρίσιμη δέσμευση και περισσότερο είναι το κρίσιμο στοιχείο και όχι η δέσμευση που έχει σημασία. Και εδώ έχουμε κυρώσει και κυρώσει των ΗΠΑ αλλά και κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάβλους επικοινωνίας οι οποίοι παραμένουν ακόμα ανοιχτοί. Αυτή η πολιτική της κρίσιμης δέσμευσης είναι αυτό, δεν είναι αυτός σκοπός. Θέλουμε να έχουμε ε, πλήρη ε, δυνατότητα και ε, μη αναστρέψιμη ε, διαδικασία παροπλισμού από, τις, από τη Βόρεια Κορέα. Επαναλαμβάνω, θέλουμε να έχουμε πλήρη ε, μη αναστρέψιμη ε, δυνατότητα παροπλισμού και των πυρηνικών και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής ε, και να μπορούμε να το επαληθεύσουμε και αυτό θα πρέπει να αφορά και τα προγράμματα βαλιστικών πυράβλων όλων των εκτάσεων και θέλουμε να μειώσουμε και τις εντάσεις στην ε, ε, χερσόνησο της Κορέας και στην ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε να έχουμε ένα παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης και έχει αναφερθεί και πόσο σημαντικό είναι αυτό νωρίτερα. Και επίση θέλουμε να βοηθήσουμε ε, να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να έχουμε μόνο διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι διαπραγματεύσεις και περιλαμβάνουν και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Βόρειας Κορέας και των ΗΠΑ καταρχάς. Επίσης να πω ότι εμείς υποστηρίζουμε τον ηγετικό ρόλο της Δημοκρατίας της Κορέας ε, και τις προσπάθειες που κάνει η χώρα αυτή να ε, διευρύνει την ε, προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών, Νότια και Βόρεια Κορέα, που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επίλυση του θέματο. Αν δεν υπάρξει πρόοδο για την αποπυρηνικοποίηση, που είναι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε δυστυχώ, θα πρέπει να πιέσουμε τη Βόρεια Κορέα μέσω κυρώσεων, να παραμείνει αυτό για να μπορέσουμε να προλιάνουμε το έδαφος για μια διπλωματική λύση. Αυτή είναι η θέση μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταφέρει όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας αμέσως και επίσης ενέκρινε περαιτέρω ε, κυρώσεις ε, μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να επιμείνουμε για την εφαρμογή αυτών των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και έγιναν και πολλές ε, ε, διαδικασίες, είχαμε διαβήματα σε τρίτες χώρες και της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας για να επιμείνουμε για την πλήρη εφαρμογή αυτών των κυρώσεων από όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι όσον αφορά τις πιέσεις. Πιέσουμε μέσω κυρώσεων. Αλλά όπως σας είπα, έχουμε και διάβλους επικοινωνίας. Και θα με ρωτήσετε πού γίνεται η επικοινωνία και νομίζω ότι ακούστηκε ήδη, δεν υπάρχει πολιτικός διάλογος σε αυτό το επίπεδο. Και θα ήθελα να σας πω σαφώς ότι αυτή τη στιγμή μεταξύ των κρατών μελών δεν υπάρχει απαραίτητη συνένεση για αυτό τον πολιτικό διάλογο και την έναρξή του. Ε, πρέπει να υπάρχει απαραίτητη συνένεση που ε, είναι αυτή η οποία οφθεί τις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές. Δεν υπάρχει συνένεση λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτικός διάλογος, αλλά υπάρχει κάποια επικοινωνία μέσω των διπλωματικών αποστολών κάποιων κρατών ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, έχουν αποστολές ε, στην Pyongyang η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Γερμανία και η Σουηδία. Είναι οι έξι χώρε που έχουν διπλωματικέ αποστολέ στη χώρα αυτή. Μέχρι πρόσφατα είχε και το Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια ω κράτο μέλο, αλλά τώρα αποχώρησε. Επομένω έχουμε έξι κράτη-μέλη με διπλωματικέ αποστολέ εκεί και η Γαλλία έχει ένα ε, πολιτιστικό γραφείο. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες επαφές με την ηγεσία της Βόρειας Κορέας, αλλά θα έλεγα ότι με πάσα ειλικρίνεια δεν υπάρχει κάποια αυθεντική πρόοδος από πλευράς Βόρειας Κορέας για έναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, ελάχιστα μπορούμε να κάνουμε εμείς και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να αναφέρω ότι κάποια πράγματα γίνονται και μέσω των διπλωματικών αποστολών που έχει ε, η Βόρεια Κορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο. Αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα. Ε, θα δούμε βέβαια τι θα αποφασίσει η Βόρεια Κορέα λόγω Brexit, διότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάει σε κάποια άλλη αποστολή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διπλωματική αποστολή δηλαδή της Βόρειας Κορέας, για περιστασιακές επαφές με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όσον αφορά τη δική μας τη δέσμευση, πρέπει να πω ότι εμείς έχουμε παρουσία μέσω περιορισμένη συνδρομής που παρέχουμε. Έχει άμεση σχέση με ανθρωπιστική συνδρομή, κυρίως είναι ε, αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά αν το δούμε και λίγο πιο λογικά, είναι ανθρωπιστική βοήθεια παρέχουμε ε, εργαλεία στους Βορειοκορεάτες ώστε να μπορούν να ε, παράγουν τρόφιμα. Αφορά την επιστημιστική ασφάλεια δηλαδή, ένα πρόγραμμα επιστημιστικής ασφάλειας το οποίο ε, είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται προς το παρόν. Δεν υπάρχει καμία ανθρωπιστική βοήθεια που εφαρμόζεται με την τεχνική έννοια του όρου από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε ξανά και ίσως είναι και μια ευκαιρία για να εξετάσουμε εάν και εφόσον θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα μέσα ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, και πάλι επίσης να πω, το είπα και στην αρχή, θέλουμε να προωθήσουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα. Η κατάσταση είναι ζωφερή, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, αλλά όποια έκθεση και αν δείτε, πρόκειται για μια κατάσταση. Ε, πολύ αυστηρές ε, ποινές φυλάκισης ή και θανατική ποινή για όσους προσπαθούν να διαφύγουν από τη χώρα. Και φυσικά εμείς προσπαθούμε με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, σε διεθνή βήματα, σε πλαίσια Ηνωμένων Εθνών, να συνεχίσουμε να πιέζουμε τη Βόρεια Κορέα, ώστε να λάβει σοβαρά υπόψη της τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δεύτερο τώρα, και θα είμαι σύντομος γιατί τα βασικά τα ακούσαμε, Ποιε είναι οι προοπτικές αποπυρηνικοποίησης τη χερσονήσου τη κορέα. Για να είμαι ειλικρινή, συμφωνώ με τα όσα ακούστηκαν. Οι ελπίδε για πρόοδο στο εγγύ μέλλον για αποπυρηνικοποίηση είναι πάρα πολύ ισχνέ. Έχουμε δει να γίνονται αρκετέ σύλλογοι κορυφή και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βόρεια Κορέα, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδο για αποπυρηνικοποίηση μέχρι τώρα. Και Υπάρχουν ε, βεβαίω ε, στι συναντήσει μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας ε, μεγάλες διαφορές για πολλά θέματα και όσον αφορά τον ορισμό του τι σημαίνει αποπυρηνικοποίηση. Εν τω μεταξύ, βεβαίως, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει τις προσπάθειές της να αναπτύξει όπλα μαζικής καταστροφής, δεν το κρύβουν. Ε, επομένως, υποθέτουμε το γεγονό ότι δεν ε, εκτοξεύουν πυράβλους για δοκιμές, ε, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε και η ανάπτυξη όπλων. Ίσα ίσα θα πρέπει να συνεχίσουμε να θεωρούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτές οι δραστηριότητε. Πότε πότε γίνονται κάποιες δοκιμές, κυρίως για βαλιστικούς πυράβλους και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι από το 2019 και μετά έγιναν περισσότερες δοκιμές βαλιστικών πυράβλων από τον Kim jong Ουλ από ότι σε όλη τη διάρκεια της ε, ε ηγεσία του πατέρα του. Ε, αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, πόρισμα. Έχουμε δει Επιτάχυση λοιπόν στις δοκιμές ε, βαλιστικών πυράβλων. Τώρα, αυτό που θέλουμε βεβαίως είναι να ξαναρχίσουν ή τουλάχιστον να υπάρξει μια ε, αυθεντική πρόοδος ε, διαπραγματεύσεων μεταξύ Βόρεια Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Παρά τι συνόδους κορυφή, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάποια σοβαρή συζήτηση σε επίπεδο εργασία για το τι θα μπορούσε να είναι από πυρηνικοποίηση. Αυτό επιθυμούμε εμεί. Αλλά δεν βλέπουμε αμέσω και αυτό φυσικά είναι ε, ε, λυπηρό και θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, κάποια προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να κάνει κάποια αποφασιστική συνδρομή για να προχωρήσει αυτή η διαπραγμάτευση. Προφανώς και ε, είμαστε σε επαφή με όλους τους ενδιαφερομένους, με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε στενές επαφές επίσης και με την ε, Νότια Κορέα που είναι στρατηγικός εταίρος όπως και η Ιαπωνία που είναι και άλλη χώρα της περιοχής που ανησυχεί και καλά κάνει για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας και τις ε, πυραυλικές δραστηριότητες. Είμαστε σε στενή επαφή με όλους αυτούς τους εταίρους, αλλά εμείς από, τους, ε, ε, από την πλευρά μας δεν έχουμε καταφέρει σε συνεργασία με άλλους να προχωρήσουμε. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και εμείς όλοι μαζί επιθυμούμε να προχωρήσει η διαδικασία, ακόμα όμως δεν έχει υπάρξει κάτι και δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια προοπτική να συμβεί κάτι τέτοιο Κυρίως λαμβάνοντας υπόψη και ότι ε, θα έχουμε προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ. κάτι φυσικά το οποίο έχει και αντίκτυπο στους ε, υπολογισμούς του Kim Κουλ. Θα πρέπει δηλαδή, εάν ε, σε αυτή την προεκλογική διαδικασία ε, θα ήταν λογικό να κάνει κάτι προκλητικό. Κατά πάσα πιθανότητα όχι. Ε, α, λοιπόν ότι δυστυχώς Έχουμε μια συνεχή κατάσταση στασιμότητας και θα συνεχιστεί αυτό μέχρι να τελειώσουν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και να είναι σαφές ποιος θα είναι πρόεδρος στο τέλος του έτους ε, ε, στις ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι τόσο συχαστικά ίσως όσα μας είπατε, αλλά πολύ ε, συγκεκριμένα και πολύ απαραίτητα και χρήσιμα. Ο κύριος Μίξερ έχει ζητήσει το λόγο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, ομιλίες τους. Ένα σχόλιο και δύο ερωτήσεις. Είναι ένα παράδοξο αυτό που βιώνουμε. Είπατε κι εσείς ότι τελικά ο απότατος στόχος του Κιμ είναι να επιβιώσει το καθεστώς του. Και ό,τι άλλο κάνει ή θέλει να πετύχει από αυτή τη βάση, από αυτή την αφετήρια ξεκινάει. Και βέβαια, αυτό το οποίο εμείς θα ήμασταν ίσως διατεθειμένοι να δώσουμε ως κίνητρο για την αποπυρηνικοποίηση, μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ της αλλαγής και όχι τόσο υπέρ της διατήρησης του καθεστώτος. Δεν θα μπορούσε το καθεστώς δηλαδή να επιβιώσει μια επαναστατική αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Αυτό εννοώ. Άρα νομίζω ότι είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να τετραγωνιστεί αυτός ο κύκλος. Και έρχομαι στις δύο ερωτήσεις μου. Τρεις μαγικές λέξεις που είπατε ήταν ότι η αποπυρηνικοποίηση θα πρέπει να είναι ε, κάτι που θα είναι πλήρες, ε, αξιόπιστο και αμετάκλητο. Είπα Νομίζω ότι επιφυλάσσονται και δεν θέλουν άρση κυρώσεων πριν πληρωθούν όλα τα κριτήρια αυτά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ή αποπυρηνικοποίησανε μετάκλητη άνευ επιστροφής πότε θα θεωρείτε Γιατί από που υπάρχει τεχνογνωσία και τεχνολογία, πάντα θα υπάρχει επιστροφή. Αλλά για να έρθουν οι, η οι κυρώσεις, πώς θα αξιολογηθεί αυτό το κριτήριο. Και για τον ενδοκορατικό διάλογο και τις ειρηνευτικές προσπάθειες τα ακούσαμε. Υπάρχουν και συνομιλίες μεταξύ Βορείας Κορέας ε, και είπα για την αποπυρηνικοποίηση. Η Ιαπωνία επίσης έχει πέσει στο τραπέζι, αλλά για την Κίνα δεν άκουσα τίποτα. Εσείς πώς θα περιγράφατε την πολιτική προσέγγιση και το ρόλο της Κίνας στην αποπυρηνικοποίηση. Ευχαριστώ, πρόεδρος Κύριε Καλνιέτη, από το ΕΛΚ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση για τις τεράστιες παράνομες ροές χρημάτων που εισραίουν στο καθεστώς που χρησιμοποιούνται και για το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά και για την κάλυψη ασδήποτε άλλης ανάγκης και για την δημιουργία της εικόνας μιας σύγχρονης πρωτεύουσα της Pyongyang Έχετε τεράστια έργα, κατασκευαστικά υποδομές, ε, οικοδομές και όλα τα άλλα ε, που γίνονται αν τα συγκρίνει κανείς με την κατάσταση στην υπόλοιπη Βόρειο Κορέα. Ευχαριστώ. Κύριε Φωτίγκα, για τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, παρέμβαση αυτή. Σημερίζομαι ε, την άποψή σας ότι πολύ λίγες είναι οι προοπτικές επιτυχίας ε, της, ε, της αποπυρηνικοποίησης τουλάχιστον σε έναν προβλέψιμο χρονικό ορίζοντα. Και εγώ ε, θέλω, όπως και προηγούμενος να αναφερθώ στην Κίνα. Η Κίνα είναι πολύ σημαντική χώρα. Έχει πολλά και διαφορετικά εργαλεία που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να υπάρξει μια θετική στροφή ή μεταστροφή της ε, Βόρειας Κορέας και το δεύτερο έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Η Βόρεια Κορέα είναι μια χώρα που ουσιαστικά δεν έχει καν σύστημα υγείας, δεν έχει υγειονομική περίθαλψη. Οι περισσότεροι στη χώρα υποσυτίζονται και μέχρι τώρα δεν έχουμε καν στοιχεία για τον κίνδυνο Ε, τι θα προκύψει εκεί αν ε, υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση. Πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Μπορεί να μην είναι ακριβώς ε, το θέμα μας στο πλαίσιο της συζήτηση που κάνουμε για την αποπυρηνικοποίηση, αλλά υπάρχει ανθρωπιστική κρίση και αν επεκταθεί, τι δυναμική θα υπάρχει εκεί. Θα είναι τελείως διαφορετική. Ευχαριστώ να απαντήσει παρακαλώ οι ομιλητές του πάνελ. Thank you very much uh, um, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις, Λέω ο Πατσέκο Πάρδο. Για το Για το πώς είναι αμετάκλητο κάτι πράγματι να κλείσουν όλες οι καταστάσεις, ε, να τους βάλεις όλους τους επιστήμονες ε, σε ένα φράκτη μέσα, να τους κλείσεις, ναι, τότε ναι, θα μπορούσαμε ότι δεν μιλάμε για επιστροφή. Ε, τώρα από την αμερικανική πλευρά το ενδιαφέρον είναι ότι τουλάχιστον κατηδίαν αλλά ίσως και δημοσία δεν γίνεται πια λόγος για τον έλεγχο όπλων κτλ ή για το πρόγραμμα αν υπάρχει επιστροφή ή όχι. Δεν ξέρω αν θα γίνει σε πέντε χρόνια, αλλά ρεαλιστικά δεν νομίζουμε ότι θα έχουμε άμεσα κάποια εξέλιξη. Και πράγματι υπάρχει στασιμότητα ε, τώρα, ε, μια τελμάτωση ε, στις επαφές μεταξύ Βόρειας Κορέας και ΗΠΑ, αλλά έχει γίνει πιο ρεαλιστική η συζήτηση και από τις δύο πλευρές. Τώρα, αν η διεθνή κοινότητα και σε ποιο βαθμό μπορεί ε, να παράσχει κάποια ανακούφιση, τέλο πάντων να άρει κάποιε κυρώσει. Άρση κυρώσεων, άπαξ και αρθούν, πώ θα τι επαναφέρει. Δεν ξέρω αν θα συμφωνούσε η Κίνα και η Ρωσία σε αυτό, αλλά το θέμα είναι να δούμε αν εκπληρώσετε τι δεσμεύσει τη ή τι υποχρεώσει τη η Κορέα, ε, θα μπορούσε να υπάρξει μια ε, ανακούφιση, ε, ένας μετριασμός των κυρώσεων κτλ. Αλλά το λεγόμενο irreversible, το κάτι που δεν έχει επιστροφή, το αμετάκλητο δεν ισχύει. Και αν δείτε το νομικό πλαίσιο στη ΣΥΠΑ δεν άλλαξε κάτι, απλά λίγο η αφήγηση, η γλώσσα που χρησιμοποιείται για το διεθνή ρόλο. Οι σχέσεις μεταξύ Βόρειας Κορέας και Κίνας ε, δεν είναι και τόσο καλές ε, από πολιτικής πλευράς, ε, αλλά χρειάζεται μια χώρα την άλλη. Ο ρόλος της Κίνας είναι κάτι πολύ σημαντικός και για λόγους συντομίας δεν αναφέρθηκα. Σι και ε, Κιμ δεν τα πάνε και πολύ καλά προσωπικά, ε, δεν θέλουν να συναντηθούν, αλλά η μόνη πλευρά νομίζω που φορά που άκουσα ε, για προθυμία της Κίνας να κάνει κάτι είναι αν θα την έπαιρνε την πυρηνική ομπρέλα που έχει τη θωράκιση αυτή η Αμερική από την Κορεατική Χερσόνησο και την πήγαινε κάποιο μακριά. Επί της αρχής, επισήμως τουλάχιστον, η Κίνα συμφωνεί για την αποπυρηνικοποίηση. Αυτό είναι ένα στοιχείο, πρέπει να το έχουν ποψή. Η Βόρεια Κορέα, Κορέα όμως έχει ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Σε βάρος της δημόσιας έρευνας ε, της ε, Κίνας. Έχουν πει πολλές φορές οι Κινές, μην κάνετε πυρηνική δοκιμή και το κάναν τη μέρα που ο Πρωθυπουργό Σάμπ είχε πάει εκείνη τη μέρα επίσκεψη, βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη. Άρα ουσιαστικά δημιουργούνται τα κίνητρα που ίσως πρόξουν την Κίνα να πιέσει την ε, Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει τα πυρηνικά. Άλλοι τέσσερι, ε, τα τέσσερα άλλα μέλη τη αντιπροσωπεία είπαν όμω ότι είναι επικοδομητική η Βόρεια Κορέα. Τώρα, κάποια άλλα ερωτήματα για τα νομικά ε, και τις παράνομες ροές χρηματοδότησης. Ε, κοιτάξτε, αν πάμε πίσω στο 2006, είχαν επιβληθεί κάποιες κυρώσεις που, από τη ΣΥΠΑ που ε, αφορούσαν μια τράπεζα μέτρα το Μακάο, επηρεάστηκε ε, η Κορέα. Είχαμε και τις συμφωνίες ε, το 2005. Ένα χρόνο ολόκληρο η Κορέα έλεγε ότι δεν κατέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν από την τράπεζα αυτή δεν αρθούν οι, κυρά, οι κυρώσεις για ένα χρόνο. Έκτοτε έχει γίνει πιο ευφύ η Βόρεια Κορέα. Ξέρει ότι μπορεί να στοχεύουν πλέον, είπα, τράπεζες που συναλλάσσονται μαζί τους σε Σιγκαπούρη, στην Κίνα και ίσως και στη Ρωσία, από ό,τι φαίνεται, ε, στη, στην Ανατολική Ρωσία. Και κάτι που βοήθησε σε κάποιο βαθμό είναι η πρωτοβουλία για την ασφάλεια και τη ε, μη, διάσωση. Κάποιες ε, ε αποστολές και καταστροφής ε, διακόπηκαν και αυτό πράγματι μπορεί να βοηθήσει. Αλλά η Βόρειος Κορέα σίγουρα είναι αρκετά μπροστά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχουν σκάρι στην Κεντρική Τράπεζα του Μπαγκλαντές και σε άλλες τράπεζες και στην Ιρλανδία και κάποιες Ιρλανδικές εταιρείες και πήραν χρηματοδότηση με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι κάπως αρνητικό. Αυτό που ίσως δεν αλλάζει τόσο είναι ότι αν μια χώρα είναι πλέον πιο ενταγμένη στη διεθνή κοινότητα, ίσως δεν έχει πλέον τέτοιες πυρηνικές βλέψεις, αλλά αυτό είναι πιο μακριά, μακρινή πιθανότητα για ε, τον κορονοϊό και αυτά που και ο κύριος Μπρέντ υπήρξε ε, η επιδημία και έκλεισαν τελείω τα σύνορα τη Βόρεια Κορέα και για τουρίστε κτλ. Και, και ότι οι διπλωμάτε μπορούν να πάνε να φύγουν από τη χώρα. Και αυτό είναι ένα ακόμη λόγο για του οποίου οι συζητήσει με τη ΣΥΠΑ θα επαναληφθούν πολύ αργότερα. Όχι μόνο λόγω των εκλογών, αλλά και γιατί φοβάται η Βόρεια Κορέα ακριβώ αυτό που είπατε, επειδή έχουν πάρα πολύ κακό σύστημα υγεία αν υπάρξει επιδημία. Πάντω, η Βόρεια Κορέα στράφηκε στη ΣΥΠΑ και ζήτησε άρση για να μπορέσει να έχει ιατρικό εξοπλισμό στη χώρα. Ίσως και κάποιοι γιατροί, αν πρόθουν να πάνε στην Βόρεια Κορέα να αντιμετωπιστεί εκεί ο κορονοϊός. Άρα εδώ ανοίγει μια ευκαιρία, ένα παράθυρο ευκαιρίας. Λέει όμως και κάτι ακόμη αυτό. Ότι η Βόρεια Κορέα μπορεί και να μην θέλει, αλλά όπως στην προηγούμενη περίπτωση χρειάστηκε να το κάνει, ίσως υπάρξουν και άλλες ε, ευκαιρίες ε, συνεργασίας με τη διεθνή κοινότητα. Και επειδή μιλήσαμε για κυρώσεις, αλλά όχι ε, έτσι, αναλυτικά, ανεξαρτήτως το αν είναι ηθικό ή όχι, ε, σίγουρα επηρεάζεται και θίγεται ο πληθυσμό της χώρας, αλλά δεν μπαίνω στο ηθικό στοιχείο. Το θέμα είναι ότι από πολιτικής και διπλωματικής, ε, αλλά και οικονομικής πλευράς, έχουν κάνει κάτι, γιατί δεν θα ζήτα για ανακούφιση ή άρση των κυρώσεων η Βόρειος Κορέα. το πρώτο πράγμα που ζητάνε από τη ΣΥΠΑ είναι αυτό, άρση κυρώσεων. Άρα ε, βλέπουμε και με την περίπτωση του κορονοϊού, όταν πλήττεται η Βόρεια Κορέα, ότι κάνει μια, έτσι, ένα άνοιγμα προς την εθνική κοινότητα. Κύριος Μπρέντερ. Ευχαριστώ. Κάποια συμπληρωματικά σχόλια τώρα. Όσον αφορά το αμετάκλητο και τι σημαίνει αυτό. Ε, στην ουσία, οι Ηνωμένε ε, και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αυτέ που μετράνε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει άποψη ένα, αλλά ο διαπραγματευτή είναι αυτό που κάνει την ερμηνεία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν θέλουν να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει μια διαδικασία καθοδόν ε, την οποία δεν θα ε, καταλάβει άλλη πλευρά. Θέλουν να ξέρουν δηλαδή ότι θα κάνουν κάποιες παραχωρήσεις ε, και δεν θα τις ε, βάλουν στο τσεπάκι τους μετά και δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα το δεχτούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αν καταλαβαίνω καλά, λοιπόν, οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν τουλάχιστον να έχουν ένα σαφή χάρτη πορεία. Θέλουν μια συμφωνία και αυτή είναι ενδιαφέρουσα ιδέα. Θέλουν μια συμφωνία με τη Βόρεια Κορέα για το πώ θα πάνε από το Α στο Β. Και το Β είναι πολύ δύσκολο να το καθορίσει ο καθένα. Τι σημαίνει από πυρηνοκοποίηση, ποιε είναι οι εγκαταστάσει. Ε, ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε και τι εγκαταστάσει του και πρέπει να μα πούνε τι έχουν, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι φυσικά να μα το πούνε και αυτό ε, για ευνόητου λόγου. Ε, είναι λοιπόν πολύ εύκολο. Αμετάκλητο σημαίνει ότι δεν επιθυμεί να δεσμευτεί η ε, πλευρά των ΗΠΑ σε μια διαδικασία που δεν είναι σαφώς καθορισμένη και δεν είναι σαφές ποιο θα κάνει τι, πότε, σε με αντάλλαγμα τι. Ε, πρέπει να ορίσουμε λοιπόν σαφώς τη διαδικασία και εξ όσων αντιλαμβάνομαι εγώ, εάν και εφόσον υπάρξουν ε, ε, εγγύησει, και θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν εγγύησει ότι μπορεί να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί ο χάρτη πορεία, τότε μπορεί να επανεξετάσουν και τη μερική άρση κυρώσεων οι ΗΠΑ. Τουλάχιστον εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι την κατάσταση. Επίσης, ήθελα να πω για το θέμα της παράνομης εισρωής χρημάτων στη Βόρεια Κορέα. Αυτό είναι θέμα μεγάλης ανησυχίας. Όντως εισραίουν χρήματα στη χώρα και η πιο σημαντική πληροφορία που έχουμε εμείς για την παρακολούθηση των χρημάτων είναι οι εκτάσει του πάνελ των εμπειρογνωμένων τη Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται συγκεκριμένα με τι κυρώσει τη Βόρεια Κορέα. Υπάρχει συγκεκριμένο φορέα λοιπόν στα Ηνωμένα Έθνη που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και έχουν ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων, διεθνών εμπειρογνωμόνων που έχουν ορίσει διάφορε κυβερνήσει και παρακολουθούν το θέμα αυτό με πάσα λεπτομέρεια και θα ρωτήσετε πώς το κάνουν αυτό βάσει εκθέσεων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών. Δεν λέω ότι έχουν την πλήρη εικόνα. Καταλαβαίνετε τι, πόσο δύσκολο είναι αυτό. Βασίζονται σε εκθέσει άλλων. Οι χώρε έχουν συμφέροντα, μπορούν και να μην μπουν απόλυτα ειλικρινώ τι συμβαίνει. Αλλά μπορεί κανεί να δει τι εκθέσει αυτέ, να τι διαβάσει. Δημοσιεύονται τακτικά, υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και δίνουν πολύ ουσιαστικέ πληροφορίες. Εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση, στα διαβήματα που κάνουμε προ τρίτε χώρε, βασιζόμαστε σε αυτές τις εκθέσεις, γιατί είναι η βασική πληρο... πηγή πληροφοριών μα, διότι δεν έχουμε ανεξάρτητε πληροφορίε για το τι συμβαίνει στι διάφορε χώρε όσον αφορά πιθανή παραβίαση των κυρώσεων. Οι εκθέσει αυτέ είναι πολύ σημαντικέ και επιτρέπουν να έχετε μια σαφή εικόνα για το πώ φτάνουν τα χρήματα στη Βόρεια Κορέα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και μέσα και επικεντρώθηκαν πολύ και σε θέματα ε, κυβερνοδιαστήματος γιατί υπάρχουν εξαιρετικές δυνατότητες. Το καθεστώ της Βόρειας Κορίας γεννά χρήματα μέσω ε, πώλησης ε, θεμάτων ε, κυβερνοασφάλειας. Η Κίνα ε, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερα. Η χώρα αυτή είναι πάρα πολύ ουσιαστική για το πώς θα μπορούσαν να κινηθούν τα πράγματα, μπορεί να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Εάν η Κίνα σοβαρά θέλει να πιέσει τη Βόρεια Κορέα, τότε θα υπάρξουν πιέσει. διότι ό,τι και γίνεται ε, σε επίπεδο εμπορίου με την ε, Βόρεια Κορέα γίνονται μέσω Κίνας. Οποιαδήποτε εμπορικά προϊόντα φτάνουν στη ε, Βόρεια Κορέα είναι μέσω Κίνα αυτή τη στιγμή. Αν θέλει η Κίνα λοιπόν να σταματήσει το εμπόριο, μπορεί να το σταματήσει και τότε η Βόρεια Κορέα θα υποστεί τεράστια πίεση. Αλλά η Κίνα δεν θέλει να λάβει σοβαρά υπόψη το θέμα των κυρώσεων, τότε τα θέματα θα είναι προ την άλλη κατεύθυνση. Η Βόρεια Κορέα θα παίρνει του πόρου που επιθυμεί. τι θα κάνουμε με την Κίνα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι the very harsh sanctions which are imposed on, on DPRK. Η Κίνα έχει εγκρίνει τις πολύ αυστηρές κυρώσεις. Η Κίνα δεν επιθυμεί να δεχτεί πυρηνικά όπλα, να δοκιμάζονται σε πυρηνικές δοκιμές στην δική της αυλή, στο δικό της χώρο. Δεν θέλει δεν μπορεί να συνομιλήσει με την Βόρεια Κορέα. αλλά θα μπορούσε να είναι ε, επικοδομητική εάν συμπεριφερθεί καλά η Βόρειο Κορέα, το οποίο τι σημαίνει όχι πυρηνικέ δοκιμέ. Ο κοροναϊός αυτή τη στιγμή πιέζει τρομερά οικονομικά την ε, Βόρεια Κορέα, ε, όπως πιέζει και άλλες χώρες, κυρίως την λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Σας ε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, σας πίεσα λιγάκι χρονικά, αλλά καθυστερήσαμε και έχουμε και ένα τελευταίο σημείο στη μερίσια διάταξη, το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών.